να αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό καταψήφισα την έκθεση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Στα πρακτικά της, τα πρακτικά θα υποβληθούν προσέγγιση του Κοινοβουλίου αρχές της επόμενη συνόδου. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσει, ήδη θα αποστείλω τα ψήφισμα τα, να καταχωρηθούν. Διακόπτεται η σύνοδος και καλό τέλος εβδομάδος σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.